για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας. High Representative, Vice President Catherine Ash... Θα ήθελα να παρακαλέσω την Πρόεδρο πρόσωπο να πάρει το λόγο. Mr. President, thank you very much. Honorable members. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί βουλευτές, ε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες των βουλευτών όσον αφορά τις πρόσφατες βιαιότητες κατά των μειονοτήτων των θρησκευτικών. 6 Ιανουαρίου εξέφρασα την τοποθέτησή μου όταν πήγα στη Βίτλεμ ε, παραμονή των, του των Ορθόδοξων Χριστουγέννων. Υπογράμμισα εκεί ότι όλες οι θρησκευτικές θρησκευτικές ομάδες πρέπει να μπορούν να συγκεντρώνονται και να λατρεύουν το Θεό τους ελεύθερα. Επίσης, καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε αμυσαλλοδοξία και κάθε βία κατά της πίστης, οποιασδήποτε και αν είναι αυτή. Κατα... Πιο πρόσφατα καταδίκασα επίσης τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο και στο Πουντζάπ. Αυτές οι επιθέσεις είναι απαράδεκτες. Διεπράχθηκαν από ακραία στοιχεία μισαλόδοξα και πρέπει πραγματικά να αντασταθούμε σε τέτοιες πράξεις. Στο σημερινό κόσμο τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται συχνά λόγω θρησκείας ή υπεπιθύσεων. Τα θύματα δεν ανήκουν σε μία θρησκεία ή σε μία περιοχή. Κάθε περιοχή του κόσμου έχει αυτό το πρόβλημα οποιασδήποτε διακρίσεις, οποιαδήποτε βία κατά ενός ατόμου λόγω των θρησκευτικών του πεπιθήσεων παραβιάζει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε παραβίαση πρέπει να εκλαμβάνεται σοβαρότατα. Η κάθε μία πρέπει να καταδικάζεται με την ίδια δύναμη και στεναρότητα, οπουδήποτε και αν λαμβάνει χώρα και οποιοδήποτε και είναι το θύμα, διότι όπως ξέρουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια χριστιανικές κοινότητες στην Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα ενώ είναι εγκατεστημένες εκεί παραδοσιακά και εναγκάζονται να μετεγκατασταθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα παραμείνει αδρανής. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους σαν πολίτες οποιοδήποτε χώρα. Ελευθερία συνείδησης ανήκει σε όλους. Ελευθερία λατρείας επίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προωθήσει τη συνεργασία της με κυβερνήσεις για να καταπολεμήσει αυτές τις πράξεις βίας και δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα των τρομοκρατών. Δεν πρέπει να δεχθούμε η θρησκεία να γίνει στοιχείο που χωρίζει τους ανθρώπους. Έχουμε παγκόσμια πρότυμα ελευθερίας, της θρησκείας και των πεπιθήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κινητήρια δύναμη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το ψήφισμα εξάλληψης όλων των παραβιάσεων αυτού του τύπου. Ομόφωνα έγινε, ε, εγκρίθηκε αυτή, αυτό το ψήφισμα το Δεκέμβριο. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να επιτύχουμε συνένεση ώστε η διεθνής κοινότητα να περάσει ένα σταθερό μήνυμα. Επίσης, εξετάζουμε μια πρωτοβουλία για να επιτύχουμε συνασπισμό δυνάμεων για το Μάρτιο πάλι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Παροτρύνουμε λοιπόν τις χώρες να εξαλείψουν τις διακρίσεις και την έλλειψη ανοχής. Οι αντιπροσωπείες μας παρακολουθούν αυτό το θέμα παντού ανά τον κόσμο και η έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ασχοληθεί με τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων ανά τον κόσμο. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το θέμα σε προτεραιότητα στην ατζέντα, μου, ατζέντα μας. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα για να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ελευθερία, τη θρησκευτική. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Βαρόνι, Άστον. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε σε αυτό το θέμα. Στο νέο έτος, στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να συζητήσουμε προσωπικά μαζί σας θέματα σημαντικά για την εξωτερική πολιτική. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Ε, εκ μέρους του ΕΛΚ ο συνάδελφος Έλμαρ Μπρόκ. Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπα, αντιπρόεδρε, κύριε πρόεδρε. Η κυρία Αντιπρόεδρος μας είπε ότι θα έρχεται πιο συχνά τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για εσά, βέβαια και για όλους του άλλου. είναι σημαντικό να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ευρεία πλειοψηφία για το θέμα αυτό και αυτό είναι νομίζω απόδειξη ότι θέλουμε να μην αρκεστούμε σε ένα απλό ψήφισμα αλλά υπάρχει κάποια άλλη συνέχεια. Έχετε δίκιο ότι η έλλειψη της ανοχής και η βία για θρησκευτικούς λόγους, άσχετα για ποια θρησκεία, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 77% των επιθέσεων που έγιναν για θρησκευτικού λόγους ήταν κατά χριστιανών. Η χριστιανική Ευρώπη θα πρέπει να αμυθεί ανά τον κόσμο, δεν επιτρέπεται να σιωπήσει. Υπάρχουν έντονες διώξεις χριστιανών όχι μόνο σε Ισλαμικές χώρες αλλά παραδείγματος και στην Κίνα και δεν θα πρέπει να δεχτούμε περαιτέρω ε, τέτοιες πράξεις γιατί η θανατική ποινή επειδή κάποιος είναι χριστιανός δεν επιτρέπεται να το δεχθούμε ότι επίσης το να παραβλέπουν οι ε, κρατικές αρχές τέτοιες ε, εκφράσεις βίας. στη Συρία, στην Τουρκία, στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Βιθλέμ και εκεί θα πάψουν πια να υπάρχουν χριστιανοί αν συνεχίσουμε τα 20 εκατομμύρια κόπτων στην Αίγυπτο βλέπω επίσης ένα πρόβλημα γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω δύο από τις απαιτήσει του ψηφίσματος καταρχήν την έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δική σας θα πρέπει να αναφέρετε το θέμα της διώξης των χριστιανών. Στην υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να έχουμε ειδικέ ε, δυνατότητες και θα πρέπει κύριε Πρόεδρε να έχουμε στις συνθήκες που συνάπτουμε με άλλες χώρες να αναφερόμαστε και στο θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας. Διακόπτε Πρόεδρο, σας ευχαριστώ εξ ονόματος Σοσιαλιστικής και Δημοκρατικής Ομάδας, ο συνάδελφος Θάνες Σβόμποντα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπετε, πρόσωπε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την σαφή σας δήλωση. Είναι πραγματικά επικίνδυνο όταν υπάρχουν όσο και περισσότερες επιθέσεις κατά των χριστιανών, όταν υπάρχει έλλειψη ανοχής στον θρησκευτικό τομέα. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το καταδικάσουμε γιατί είμαστε υπέρ της ε, θρησκευτική ανοχής και ελευθερίας. Θα πρέπει να εκφράσουμε την συμπόνια μας και τη λύπη μας για τις ε, επιθέσεις κατά των κόπτων χριστιανών στην Αίγυπτο. Αυτό ήταν μια, ένα σημαντικό πλήγμα όχι μόνο κατά των κόπτων χριστιανών αλλά και κατά της ε, ανοχής που ακόμα και τονίζω ακόμα υπάρχει στην Αίγυπτο. Επίσης λοιπόν στα πλαίσια της ομάδας μου και για αυτά που γίνονται στο Ιράκ κατά των χριστιανών δεν ήταν και αυτός ο στόχος ε, της ε, ε, πτώσης του Σαντάμ Χουσέινα υπάρχει τώρα αυτή η έλλειψη ενοχής κατά των χριστιανών. Από την άλλη μεριά υπάρχει σε άλλες χώρες και έλλειψη ενοχής έναντι άλλων θρησκευτικών ομάδων, ιδίως μειονοτήτων. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι κατά των πρακτικών αυτών. Σχεδόν, δεν κάνω ποτέ γραπτές ε, δηλώσεις, αλλά προσκλήσει του συνεδέρφου Μαωρέ το έκανα γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή την αυξανόμενη έλλειψη ανοχής και έτσι έχουμε ένα κοινό ψήφισμα, μια κοινή βάση δηλαδή δράσης. αλλά εξ ονόμα μας ομάδα μα θέλω να εκφραστώ κατά οποιασδήποτε επίθεση, όχι μόνο αυτών των αιματηρών επιθέσεων, αλλά κάθε επίθεση κατά το Και να σα πω ότι από την άλλη μεριά λυπούμε ότι υπάρχει μια Ισλαμοφοβία, αν θέλετε, όσο πάει αυξανόμενη στην Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι ένα περαιτέρω επιχείρημα που ορισμένες δυνάμεις ριζοσπαστικές των μεομεθυνών θεωρούν ότι αυτό μπορεί να δικαιολογήσει τις δικές τους επιθέσεις κατά των χριστιανών. Όλοι νομίζω, όπως και να αξιολογούμε εμείς τις διάφορες ε, θρησκείες, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν ε, την θρησκεία τους ελεύθερα, ήσυχα και υπάρχει μία μειοψηφία ανθρώπων που είναι έτοιμοι να ασκήσουν βία στους χριστιανούς, στους Ισλαμιστές, στους Εβραίους, αλλά δεν έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να μπορούν να το κάνουν αυτό. Ευχαριστώ. Πρώτα σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαριέτ Χεσχάκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε αντιπρόσωπο συνάδελφοι. Η θρησκευτική πεποίθηση είναι διαφορετική υπόθεση για το κάθε άνθρωπο. Πρέπει να έχουν την δυνατότητα του, να συναντώνται σε όλο τον κόσμο. Και εξετάζοντας τον κόσμο σήμερα τα πράγματα δεν είναι καλά από το Ιράν, την Αίγυπτο, στο Πακιστάν. Έχουμε επιθέσεις κατά των χριστιανών και στο Ιράκ και στην Ιγυρία. Σήμερα μιλάμε για την ενισχυμένη βία κατά των χριστιανών και προκαλεί μεγάλη ανησυχία αυτό. Είναι πολύ οδυνηρό να έχουμε επιθέσεις για λόγους θρησκευτικούς. Όλες οι θρησκείες είναι θύματα. ορισμένα ακραία στοιχεία επιλέγουν τη βία και την τρομοκρατία εν ονόματι του Θεού τους και ισχυρίζονται, ε, προσωπεύουν και άλλους και ότι είναι υπεράνω του νόμου. Και έτσι συνδυάζουν αυτή τη βία αναρρύθμιτους ανθρώπους δεν πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο με τους τρομοκράτες από ό,τι πρέπει. Συνδέοντας τη τρομοκρατία με τη θρησκεία, ουσιαστικά δημιουργούμε πρόβλημα για όσους θρησκεύονται. Ε, η τρομοκρατία είναι πολιτικό θέμα και είναι έγκλημα. Η θρησκεία δεν μπορεί ποτέ να είναι αξιόπιστος λόγος για τη χρήση βίας. Πολύ συχνά αυτό συμβαίνει, όχι μόνο μέσω βίας, αλλά περιορίζεται και η ελευθερία του λόγου όπως μέσω νόμων για τη βλασφημία. Ποτέ δεν πρέπει να ζουν οι άνθρωποι για τη θρησκεία τους μέσα στο φόβο. Είμαστε κατά των ακραίων πράξεων, κατά των χριστιανών και υποστηρίζουμε όσους καταδικάζουν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια. Η κυρία Νικόλ Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι ιδιότητες ε, τις οποίες ε, υπέστησαν οι κόπτες στην Αλεξάνδρεια ήταν ένα θλιβερό γεγονός. Η κατάσταση των ε, χριστιανών στην ε, Παλαιστίνη, στο ε, Λίβανο, στο Ιράν είναι τραγική. Οι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τι χώρε αυτές ταπεινωμένοι. Ε, ήθελα να σας χαρώ διότι το φύσμα για τη θρησκευτική ελευθερία υπενθυμίζει τα θεμελιώδη ζητήματα, δηλαδή το δικαίωμα στην πίστη και το δικαίωμα στην μη πίστη. Το κείμενο μας αναφέρει πολύ σωστά τις πρόσφατες ε, επιθέσεις και δολοφονίες που έγιναν απαναχού στον κόσμο. Πρέπει να δεχθούμε ότι σε ορισμένε ευρωπαϊκές χώρες ο σεβασμός αυτής της ε, σκεφτικής ελευθερίας ε, διακυβεύεται. Βλέπουμε ότι συχνά υπάρχουν βεβηλώσεις νεκροταφείων, δράσεις αντισημιτικές κλπ. Η απαγόρευση ε, ε, δημιουργίας μιναρέδων στην ε, Ελβετία δείχνει μια άνοδο της έλλειψης ανοχής. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε υπόψη τους ετούντες άσυλο, τους μετανάστες αλλά και τις θρησκευτικέ μειονότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν συχνά την παραβίαση των θεμελιών δικαιωμάτων τους. Η Ευρώπη χρειάζεται να είναι υποδειγματική σε ό,τι αφορά την ανοχή και τον διαθρησκευτικό διάλογο. Οι μουσουλμάνοι της Ευρώπης ε, συνδέονται με τον Ισλαμισμό και την τρομοκρατία συχνά, κάτι το οποίο δεν αληθεύει. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ποίημα του Λουί Ραγκό, αυτός ο οποίος πίστευε στον ουρανό, αυτός ο οποίος δεν πίστευε στον ουρανό, έχουν το ίδιο αίμα, του ίδιου χρώματος και της, την ίδιας ε, φύσης και λαμπρότητας. Το λόγο έχει ο κύριος Ζημάνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, είπα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την είπατε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για την τάχιστη αντίδρασή της τα όντα συνέβησαν στην Αλεξάνδρεια. Μόνο αν αντιδρούμε άμεσα, τότε η φωνή μα ακούεται στον κόσμο. Οι χριστιανοί είναι η μειονότητα η οποία έχει ξεχαστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. χιλιάδες ε, χριστιανοί διώκονται ανά τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τις ε, θρησκευτικέ ελευθερίες που θα πρέπει να βελτιωθούν τόσο στο Σουδάν, στο Ιράκ ε, και στο Ιράν, την Αίγυπτο και Αλαχού. Ιράν λοιπόν, Βιετνάμ, Κίνα θα πρέπει να γνωρίσουν τι σημαίνει τη θρησκευτική ελευθερία. Νομίζω ότι αυτό εμπεριέχεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουμε με τις χώρες αυτές τώρα. Σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο πρέπει να ε, ε, ε, βελτιώσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των χριστιανών. Έχουμε μέσα, έχουμε εργαλεία στη θέση δεν πρέπει να φοβηθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι η ελευθερία των χριστιανών είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για μας και θα εισακουστούμε μόνο εάν αυτό γίνει κατανοητό. Διαφορετικά δεν μπορούμε να περιμένουμε μια επιτυχή ε, εξέλιξη. Το λόγο έχει ο κύριος Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας το δικαίωμα του κάθε ατόμου να ακολουθεί την οποιαδήποτε θρησκευτική πεποίθηση ή και καμιά πρέπει να κατοχυρώνεται και να γίνεται σεβαστό από όλους. για μας δεν νοείται η θρησκεία να γίνεται εργαλείο εκμετάλλευσης σε πολιτικές συγκρούσεις. σε αυτό το πλαίσιο καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα τόσο στην αλεξάνδρεια όσο και αλλού και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων σε μια πρωτοφανή ενέργεια από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς στην κύπρο η χριστουγεννιάτικη θρησκευτική τελετή στην εκκλησία του αγίου Συνεσίου στο κατεχόμενο ριζοκάρπασο διακόπηκε βία και τελικά ακυρώθηκε παραβιάζοντας θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων όπως αυτό της θρησκευτικής ελευθερίας ενώ ομοίως στη γιαλούσα την ημέρα των θεοφανίων ακυρώθηκε με τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι η άδεια δεν είχε ληφθεί εντό του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματο. οι ανωτέρω πράξει, κύριε πρόεδρε παραβιάζουν ξεκάθαρα τη συμφωνία της Τρίτη βιέννης τη Δευτέρα αυγούστου του 1975 καθώ και το άρθρο 3 και 9 τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζουμε έντονα τις ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος οι οποίες συνιστούν κατάφορη παραβίαση ενός από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. χρειάζεται επίγουσα αντίδραση. ο σεβασμό των πεπιθήσεων και των δικαιωμάτων πρέπει να έχουν θεμελιώδη σημασία για την ευρωπαϊκή ένωση. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράκ και στην Αίγυπτο είναι εγκληματικές πράξεις που εκπροσωπούν μόνο μια πτυχή των διώξεων των χριστιανών ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Μέση Ανατολή. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο από θεσμική σκοπιά είναι ο συστηματικό περιορισμός των δικαιωμάτων των χριστιανών ως πολιτών που δεν τους επιτρέπει να οικοδομούν εκκλησίες, να έχουν πρόσβαση σε διάφορα αξιώματα αλλά και να μην έχουν δυνατότητα ελεύθερης λατρείας. Τρομοκρατία και διάκρισης οδηγούν στην ε, μετανάστευση δεκάδες χιλιάδες πολιτών στο Ιράκ πάνω από το 60% των χριστιανών υποχρώθηκαν στην, σε εξορία και μιλάμε για 600.000 άτομα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται για τα δικαιώματα των λαών να μεταναστεύουν. Σε αυτή την περίπτωση όμως ε, αρνούνται το δικαίωμα των πολιτών να ζουν στην ίδια του τη χώρα κατά της τρομοκρατίας που με τις τραγωδίες θέλει να εκδιώξει τους χριστιανούς από τις αραβικές χώρες θα πρέπει να δράσουμε με διάφορα μέσα και με στρατιωτικά. Αλλά η Ευρώπη η οποία είναι ε, μια χριστιανική επικράτεια θα πρέπει διακόπτει ο πρόεδρος ο κύριος Γκόλινς έχει το λόγο. Η ελευθερία της συνείδησης οπωσδήποτε είναι ουσιαστικότατη. Ο Θεός δεν μπορεί να θέλει υποχρεωτική προσχώρηση. Αυτή η ελευθερία διώχθηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς. Πρέπει κανείς να έχει το κουράγιο σήμερα να το πει ότι αυτές οι παραβιάσεις βασικά διαπράττονται κατά των χριστιανών σε ισλαμικές χώρες. Σωστά καταδικάζονται οι φοβερές επιθέσεις φανατικών. Δίκαια το πράττουμε. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο εξτρεμιστές. Σε πολλές χώρες Ισλαμιστικές, ακόμη και με τριοπαθείς, οι χριστιανοί είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Τιμωρούνται καμιά φορά, ακόμη και με θάνατο. Λοιπόν, η κυρία Κιλ Νίλσεν μπορεί να είναι δυσαρεστημένη, αλλά κανείς στη Δύση δεν παρεμποδίζεται να γίνει μου αμεθανώσαν αν το επιθυμεί. Οι απόπειρε. Τώρα, η νομοθεσία σε σχέση με την βλασφημία πρέπει να καταργηθεί και ζητάμε ειδικότερα το Πακιστάν να ανατρέψει την απόφαση κατά μιας γυναίκας που καταγγέλθηκε από τους γείτονες. Πρέπει να περάσουμε το σωστό λόγο στους άλλους και στις σχέσεις με τα κράτη πρέπει να τους αποσαφηνίσουμε ότι οφείλουν να έχουν σεβασμό της ελευθερίας της συνείδησης για να έχουν να αξιόπιστα τα κράτη μαζί μας. Ο κύριος Μάουρο Μάριο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για το περιεχόμενο της παρεμβάσεώς σας, διότι ο σκοπός αυτού του ψηφίσματός μας είναι να εγγυηθούμε μεγαλύτερη προστασία των ε, θρησκευτικών μειονοτήτων και αυτό προς ε, όφελος και για το καλό όλων. Θα ήθελα όμως να σας παρατηρήσω το εξής. Εάν έχετε την υπομονή να ξαναδιαβάσετε το κείμενο που μας αναγνώσατε, θα διαπιστώσετε ότι η όλη σας παρέμβαση δεν, ανέφερε, δεν περιέχει τον όρο χριστιανή. Αυτό είναι κάτι το οποίο με εξέπληξε, διότι στα θεσμικά μας όργανα υπάρχει πραγματικά μια ε, δυσαρέσκεια, διότι ε, παίζουμε με αυτόν τον τρόπο τον ε, παιχνίδι των ακραίων που θέλουν να υπάρξει κάποια σύγχυση ανάμεσα στους ε, χριστιανούς αλλά οι χριστιανοί του οι Άραβες χριστιανοί αγαπούν τις χώρες τους οι Λιβανέζοι χριστιανοί αγαπούν τη χώρα τους οι Αιγύπτιοι επίσης σας ρωτώ λοιπόν κυρία Ήπατη πρόσωπε. δεν θα πρέπει να κάνουμε μια εξέταση της συνείδησεώς μας, μια ανάλυση για να δούμε το πώς έχουμε προσεγγίσει το ζήτημα μέχρι τώρα, διότι θα πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάφη σκάφη, να είναι πράγματα με το όνομά τους θα πρέπει να ονομάζουμε το μίσος κατά των Εβραίων αντισημιτισμό, το μίσος κατά των Μουσουλμάνων Ισλαμοφοβία και το μίσος κατά των Χριστιανών με, τον, με τη σωστή ονομασία. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να, ε, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις ε, τα άτομα τα οποία ε, είναι οπαδοί της ειρήνης ε, και της ελευθερίας τώρα σε ό,τι φορά τις συμφωνίες με το Ιράκ θα πρέπει λοιπόν μέσα στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών να θέσουμε σαφείς κανόνες έτσι ώστε να υπάρξουν ε, εμπορικά ωφέλη αλλά και ελευθερίες, δικαιώματα. Ας κάνουν τα πράγματα σωστά διότι ο κόσμος περιμένει ένα μήνυμα από την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ρίτσαρτ Χόβιτ για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ε, τα λόγια της παγκόσμιας διακήρυξης. Ελευθερία, θρησκείας και λατρείας, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Η παρατήρηση είναι ότι η προστασία αυτής της ελευθερίας είναι αδύνατον να ξεχωριστεί από τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να προασπιστεί ακόμη δηλώνεται ότι θα πρέπει να είμαστε κατά οποιασδήποτε θρησκευτική δίωξη. όπου και αν εμφανιστεί. 70% των ανθρώπων ζουν σε χώρες με πολλούς θρησκευτικούς περιορισμούς. Πιστεύω ότι η θρησκεία μπορεί να είναι κινητήρια δύναμη για το καλό και προωθούμε στην περιφέρειά μου αμοιβαία κατανόηση για διάλογο όπως αυτό διατυπώνεται και στο ψήφισμα. Αλλά όταν ο Τέρι Τζόντς απειλεί το Κοράνι αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί και στη δικιά μου περιφέρεια αναστάτωση. Του είπαμε όμως ότι δεν θα γίνει δεκτός. Η ανοχή και η αμοιβαία κατανόηση προωθεί τις αξίες σωστά. Αυτές είναι αξίες που πρέπει να σεβαστούμε. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Μαχιέλ Ντοσαχνέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο φανατισμός που στοχεύει κατά μια άλλη θρησκείας είναι μια βαρβαρότητα και πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό σήμερα να είμαστε αλληλέγγυοι με όλους εκείνους που διώκονται για τη θρησκεία τους, την πίστη τους παντού οι φοβερές επιθώσεις του, της Αλκάιντε στο Ιράκ και στην Αίγυπτο και ο φονταμεταλισμός κατά των χριστιανών της Μέσης Ανατολής ουσιαστικά παροτρύνει στο μίσος, φέρνει σε αντιπαράθεση τις κοινότητες, προκαλεί ένα πολιτισμικό σοκ. Πρόκειται για προσπάθεια αποσταθεροποίησης για την Ευρώπη και για τη Γαλλία. Όλη η μουσουλμανική κοινότητα βεβαίως καταδίκωσε αυτές τις βάρβαρες πράξεις. Σήμερα πρέπει να επιβεβαιώσουμε το δικαίωμα κάθε μειονότητας να ασκεί ελεύθερα και ανασφαλεία τη θρησκεία της, οπουδήποτε στον κόσμο και βεβαίως και σε εμά στην Ευρώπη. Πρέπει να προασπίσουμε τον θρησκευτικό πλουραλισμό, την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς διατυπώνω την ευχή η δημοκρατική επανάσταση να περάσει στην Τινησία και να επεκταθεί σε άλλες χώρες ώστε να διαχέονται οι αξίες του σεβασμού, της κοσμικότητας και της ανοχής. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Ο συνάδελφος Πέτρο Βαντάλεν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άστον που βρίσκεστε ανάμεσά μας. Συχνά στο Κοινοβούλιο συζητήσαμε θέματα από αφορούν χριστιανούς στο Σουδάν, τη Σομαλία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, στο Ιράκ, στο Ιράν, στο Αφγανιστάν, τη Μαλαισία και στο Πακιστάν. Πόσες και πόσες ερωτήσεις το Κοινοβούλιο και η ομάδα μου δεν έθεσαν ε, για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες αυτές. Νομίζω ότι πέρασε ο χρόνος ε, για να κάνουμε δηλώσεις, πρέπει να περάσουμε σε δράση. Έχω δύο συγκεκριμένα θέματα να τα θίξω, κυρία Άστον. Πρώτα απ' όλα, ε, η εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να πάρει στα σοβαρά το εξής να προστατεύσει τους διακόμενους χριστιανούς. Άρα να συσταθεί μια ειδική μονάδα που θα ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διμερείς ε, σχέσεις ε, και συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Θα πρέπει να τις παγώσουμε, να τις βάλουμε στην κατάψυξη. Πρέπει να πλήξουμε αυτές τις ε, κυβερνήσεις και οικονομικά μέχρι ότου χορηγήσουν τις απαραίτητες ελευθερίες στους χριστιανούς. Επόμενος αγορητής, είναι η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, η ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς δεν ε, ε, προσυπέραψε το ψήφισμα που εξετάζουμε σήμερα. Φυσικά θα πρέπει να καταδικάσουμε όλε τι τρομοκρατικέ πράξει από όπου και αν αυτέ προέρχονται, όποια και αυτά τα θύματα και όπου και αν αυτέ διεξάγονται. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε οπαδοί του κοσμικού κράτου. Καταδικάζουμε φυσικά την ε, βλασφημία. Αλλά αυτό σημαίνει παράλληλα ότι είμαστε υπέρ τη ελευθερία τη σκέψη, τη ελευθερία συνειδήσεων και τη άνοιξη τη θρησκεία. Μπορεί κανεί να πιστεύει, να μην πιστεύει, να διαλέγει την θρησκεία του και να επιλέγει και τον τρόπο λατρείας οποιαδήποτε και αν είναι η θρησκεία του. Θα, το σημαίνει επίσης ότι είμαστε, θέλουμε να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική και την θρησκεία και καταδικάζουμε την αναζωπήρωση των ε, ακροατήτων στον θρησκευτικό τομέα στην ανά τον κόσμο. Θεωρούμε ότι αυτό το ψήφισμα δεν πηγαίνει προς την κατεύθυνση. Θα έλεγα με λίγα λόγια ότι δεν έχει την απαραίτητη ισορροπία σε σχέση με αυτή που κατέθεσε η ομάδα μου. Κατά εμά αυτό το ψήφισμα δίνει εντύπωση ότι η χριστιανική κοινότητα της Ευρώπης τρέχει για να βοηθήσει τους χριστιανούς ανά τον κόσμο. Εμεί δεν θέλουμε διακόπτη ο πρόεδρος, ο κύριος Μπέλντερ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Δικαίως αυτό το ψήφισμα αναφέρεται στη βία κατά των θρησκευτικών μενοτήτων. Ένας ε, Εβραίος φοιτητής που γνώρισα τελευταία μου είπε ότι αρχίζω και φοβάμαι, φοβάμαι πού μπορώ να πάω για να είμαι ασφαλισμένος. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι θα κάνει η Ευρώπη στο μέλλον όσον αφορά τους Εβραίους συμπολίτες μας. Το ίδιο ισχύει και για τους ε, χριστιανούς ε, στην Μέση Ανατολή. Η παλαιστινιακή μειοψηφία επίσης ε, περιμένουν να τους υποστηρίξουμε. Θα πρέπει οι χριστιανοί να φροντίσουν ε, παιδιά Παλαιστινίων με ειδικέ ανάγκες να προστατευτούν, να ενισχυθούν. Υπάρχουν προβλήματα για την καθημερινή ζωή. Υπάρχει αυτό, για να αναφερθεί, αλλά η Κομισιόν ως σημαντικός ε, χορηγός της ε, Παλαιστινικής κοινότητας πρέπει επίσης να συμμετάσχει στις προσπάθειες αυτές. Η κυρία Ντότ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω για ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ως εσένας, ε, βλέπω όσο πάει και περισσότερο η χριστιανική θρησκεία να θεωρείται απαράδεκτη σε μια κοινωνία στην οποία θα πρέπει ή να πιστεύουμε όλοι τα ίδια ή να μην πιστεύουν τίποτα. Αυτή η επίθεση πάνω στα πιστεύω είναι πάρα πολύ έντονη κατά των χριστιανών σε ορισμένε περιπτώσει. Φέτο έχουμε την 400η επέτειο τη ε, βίβλου του, ε, του Ιακώβου του King James Bible. Η, άμα σε αυτό δεν φαίνεται να μας επηρεάζει υπάρχουν ε, ε, απαγορεύσεις ορισμένων ε, επαγγελμάτων σε χριστιανούς για τη οδυσία τους ή στο Ηνωμένο Βασίλειο τη νόμη για την ισότητα κατά κάποιο τρόπο τιμωρούν την έκφραση της χριστιανικής πίστης. Αυτό απεδείχθη πρόσφατα από την Κομισιόν όταν δημοσιεύσανε το ημερολόγιο τους. όπου αναφέρονται όλες οι γιορτές, μαθηματικές, εβραϊκές, βουδιστικές και άλλες, αλλά όχι χριστιανικές γιορτές. Είμαι σίγουρη ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο και καλό την είπα το πρόσωπο να το λάβει αυτό υπόψη της στα σχολεία της. Η ελευθερία έκφρασης της θρησκείας είναι μια βασική, ένα βασικό δικαίωμα των πολιτών και θα πρέπει να μπορούν να την εκφράσουν. Δεν θα πρέπει δηλαδή να διστάσουμε να εκφραστούμε γιατί πρόκειται για ε, χριστιανούς οι οποίοι διώκονται. Ο κύριος σε δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ πρόεδρε, εξότιμη κυρία Πατακπρόσωπο, κύριε κυρία αντιπρόεδρο. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δήλωσή τη, η οποία ήταν πολύ σωστή, έγινε την κατάλληλη στιγμή. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική όσον αφορά τη βασική στάση της υπηρεσίας σας και τη δική σας σχετικά με τη συνεργασία με άλλες χώρες, σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα. Αυτή είναι μια συζήτηση που είναι απαραίτητη εδώ στο σώμα, όχι μόνο λόγω της ε, πρόσφατης ε, των προσφάτων ε, κρουσμάτων, αλλά και γιατί η έκφραση της θρησκευτικής πίστης είναι ένα τμήμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Είναι ιδιαίτερα ενσυγητικό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ε, θυμάτων των διώξεων αυτών είναι χριστιανοί. Και γι' αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας σε εκείνους που ε, σκοτώθηκαν ε, ή τραυματίστηκαν ή βασανίστηκαν μέσα στα πλαίσια αυτών των ακριοτήτων. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειωθεί αυτό. Δυστυχώς γνωρίζουμε τις διακρίσεις κατά των χριστιανών και από τις αρχές και αυτό θέλουμε να το μειώσουμε. Δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πολύ λέει πρόεδρο. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γι' αυτό χρειάζεται να δεσμευτούμε εμείς για την επικράτηση της θρησκείας Θέλουμε να το έχουμε αυτό πάντα κατά νου σε όλες τις διμερείς σχέσεις. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέσα να χρησιμοποιούμε στην περίπτωση κρίσης, στην περίπτωση της προστασίας της θρησκευτική ελευθερίας και γι' αυτό χαιρετίζουμε σε όλες τις διμερείς επαφές η επιβολή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και όσον αφορά την ανεξιθρησκεία να εφαρμόζεται. Και αυτό είναι καλό να συμπληρωθεί μια σχετική ρήτρα στι συμβάσει μα με τι τρίτε χώρε. Και χαίρομαι που θα αφιερώσετε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της αλεξιθρησκείας. Ε, ευχαριστώ Λεπρός, και με συγχωρείτε για άλλη μια φορά που σας ε, ανεστήξα. Ο κύριος Γκίνο Μιλάνα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε η καταδίκη αυτών των επιθέσεων και η αίτηση για λήψη κατεπηγόντων ε, μέτρων στον ανά κόσμο είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει φυσικά απόλυτα σύμφωνος. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που δολοφονείται σε μια εκκλησία και κάποιον ο οποίος δολοφονείται για λόγους ε, ε, απάτης ε, ή για κάποιους άλλους ε, λόγους, μοιχείας κλπ. Το δικαίωμα στην ε, ελευθερία και στην συνύπαρξη είναι κάτι το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τις διεθνείς συμβάσεις. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στους οπαδούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολέμιους αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να τηρηθούν αυτές οι ελευθερίες, κάτι το οποίο διαφορετικά οδηγεί σε έξοδο αυτών των ε, θρησκευτικών μειονοτήτων από τις χώρες του οποίες κατοίκουν. Θα πρέπει λοιπόν να λεφθούμε μέτρο από την Ευρώπη σε ε, πολιτικό και πολιτικό επίπεδο. Ζητάμε λοιπόν από την αρμόδια επίτροπο να υιοθετήσει σαφείς κατήγραμμες στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο της νέας ε, υπηρεσίας εξωτερικής πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την άνεξη θρησκεία. <clears throat> Πιστεύω μεταξύ όλων την ε, τον ε, διαψυχιακό διάλογο ο οποίος είναι απαραίτητος για να ξεπεράσουμε παρόμοιες καταστάσεις και να αποφύγουμε πολέμους οι οποίοι ξεκινούν από θρησκευτικέ ε, διαφορές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και την κατάσταση που στην Ευρώπη όπου υπάρχει έλλειψη ανοχής. Αυτό το ζούμε καθημερινά σε διάφορες περιοχές και προάστια πόλεων. Χρειάζεται λοιπόν να φροντίσουμε, να φροντίσουμε να τηρηθούν αυτές οι ελευθερίες θρησκευτικέ. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, διακόπτει ο Πρόεδρος, διαβάζεται πάρα πολύ γρήγορα και οι διαρριμνείς μας αντιμετώπιζαν προβλήματα. Ο κύριος Ρινάλντι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την είπατε εκπρόσωπο, Αγαπητή συνάδελφοι. Η κατάσταση στην ε, Μέση Ανατολή ε, τα δημιουργεί ε, κάποιες διαφοροποίησεις δεν θα πρέπει όμως να, κάνει το, τα να κάνουμε το λάθος να μιλήσουμε για συγκρούσεις πολιτισμών. Πριν από μερικά χρόνια στο Κάιρο ένας πρώην ε, Γιώργος ε, που μας έφερε το γάλα στο σπίτι μας χτύπησε την πόρτα κλαίγοντας δεν καταφύραμε τι λέγανε τι ήθελε να πει έλεγε Σαχίν Ακμπάρ ο ο ηλικιωμένος, μεγάλος ηλικιωμένος ήθελε να εκφράσει λοιπόν τον ε, θάνατο την λύπη του για το θάνατο του Πάπα Κάρολ Βολτίλα του οποίου ήταν ιδιαίτερος θαυμαστής αυτός το μικρό αλλά σημαντικό επεισόδιο το οποίο δείχνει το πώς σκέφτεται η ε, ο Αιγυπτιακός πληθυσμός συνέβη στην χώρα όπου οι κόπτες δολοφονήθηκαν πριν από τρεις εβδομάδες. Χρειάζεται λοιπόν να λάβει υπόψη της η εξωτερική πολιτική. Πρόεδρος διακόπτη, διαβάζετε και εσείς πάρα πολύ γρήγορα. Δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική θα πρέπει να μην φοβηθεί να μιλάει για την χριστιανοσύνη και για τους χριστιανούς Γι' αυτό προ όφελο των δημοκρατιών και των δημοκρατικών διαδικασιών. Ευχαριστώ, η κυρία Η κυρία Μαρίνα Γιανγκουδάκη. Ένα λεπτό. Η ενοχή, των πιστεύω των άλλων, είναι χαρακτηριστικό πολιτισμένη κοινωνία. Οι παραβάσει στην ΑΕΤΟ ε, είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικές. Ε, είτε αυτές οι επιθέσεις γίνεται κατά χριστιανών είτε άλλων ε, θρησκειών είναι απαράδεκτες στην κοινωνία αλλά πριν επικρίνουμε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε εμά. Τον περασμένο μήνα απαγορεύτηκαν στο Κάπαστο παρεμποδίστηκαν μάλλον στο Ρισοκάπαστο οι, χριστιαν... η των Χριστουγέννων. 36 χρόνια ήταν η περιοχή αυτή υπό τουρκική ε, κατοχή και το να μπουν ο στρατός στην εκκλησία και να ε, επιβάλλει στον ε, ιερέα να σταματήσει τη λειτουργία και να φύγουν οι χριστιανοί, οι πιστοί, είναι απαράδεκτο. Αυτό εξετάζεται από τον ΟΗΕ αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρώτη πρώτα να κανονίσουμε τα του οίκου μας δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία ε, τέτοια παράβαση εδώ εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Το Γιόν Κορνελής για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Ιεπατα Πρόσωπε, η ανεξηρεσία προστατεύει τις θρησκείες οι χώρες έχουν την υποχρέωση να ε, προωθήσουν την ανοχή και να προασπίσουν εκείνους που είναι θύματα διακρίσεων ή βίας. Χαιρετίζω γι' αυτό το κοινό ψήφισμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι επειδή πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με τους στενούς, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή οι χριστιανοί ε, έχουν να αντιμετωπίσουν πραγματικά έλλειξη ενοχή σε πολλές χώρες. Ακόμα και αν αυτό αφορούσε και άλλες ε, θρησκείες θα είχαν την ίδια στάση. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Εγώ είδε, είχα στο ανάλογο Ολλανδικό Υπουργείο κάποια θέση που σχετίζονται με αυτά τα θέματα και είδα πόση προσπάθεια και πόσο προσωπικό χρειάζεται για να ανεμεστούν αυτού του ίδιου τα προβλήματα και πίζω κύριε Αντιπρόεδρε, θα μπορέσετε πραγματικά να έχετε τη δυνατότητα να αντιπρόσετε το θέμα. Υπάρχει ένας όρος ταμπού, ε, χριστιανοφοβία, αλλά από πολλές πλευρές ε, εδώ και χρόνια μας φτάνουν ειδήσει ε, πολύ σοβαρές και τραγικές για τις διώξεις χριστιανών ανά τον κόσμο. Η Ευρώπη θα πρέπει να ξυπνήσει να ανοίξει τα μάτια της και να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα. Παραδείγματο χάρη αυτό το οποίο περιμένω από την κυρία Άστον είναι ότι θα μπορούσε να αναφερθεί στα λόγια του Πάπα Βενεδίκτου που ανέφερε ότι η άρνηση της σκεφτικής ελευθερίας ε, φύγει ε, τον, ε, το Θεό αλλά και την ίδια την ειρήνη. Τι περιμένει λοιπόν να στείλει αποστολή στην ε, Αίγυπτο για να δει το πώς ζουν οι κόπτες ε, οι οποίοι είναι χριστιανοί μετριοπαθείς δεν μπορούν καν ε, να αναλάβουν κάποια κάποιες θέσεις Ευρώπη ξύπνα θυμίσου τις χριστιανικές σου Ευχαριστώ κύριε Μποργκέζη επόμενος αγορητής είναι ο κύριος Μαγιόρ Ορέχα για δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε ε, επιθέσεις που προσφάτως συνέβησαν στο Ιράκ και στην Αίγυπτο δείχνουν ε, δύο τραγωδίες για την Ευρώπη αν και είναι διαφορετικής φύσης. Πρώτον τραγωδία για τα γεγονότα αυτά καθεαυτά για την ε, δολοφονία ανθρώπων αλλά είναι και τραγωδία επίσης ο τρόπος με τον οποίο περνάει στα ψηλά τέτοιο γεγονός της κοινωνίας μας Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση διότι έτσι θεωρείται ότι σαν να επρόκειτο μία επίθεση κατά κάποιων ξένων ε, ζώντων σε μακρινά σημεία του κόσμου. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά πλήττουν τον ίδιο τον πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα και το εύρος αυτών των επιθέσεων κατά των χριστιανών. Και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρειάζεται όχι μόνο να κάνουν δηλώσεις γενικόλογες και καταδίκες, χρειάζεται να αναλάβουν μία σειρά δράσεις δύο ειδών. Πρώτη δράση είναι ότι τέτοιες ε, τραγωδίες ε, δεν θα πρέπει να επαναληφθούν και να είναι να, ε, και να ενημερώνουν πιο πολύ τους πολίτες. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο Επιτρέψτε μου κυρία Αντιπρόεδρε να πω ότι ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εσείς η ίδια θα πρέπει να βοηθήσετε τα θύματα αυτών των καταστάσεων. Χρειάζεται να τρέξετε για να βοηθήσετε αυτά τα όργανα, αυτά τα άτομα. Χρειάζεται να υπάρξουν κάποιες, ε, προγράμματα συναντήσεων, επαφών, προγράμματα στήριξης ε, των θυμάτων. διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν αυτήν την φρικτή δίωξη που υφίστανται. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαυρονικόλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ως σοσιαλιστές πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα και ασφαλώς στα θρησκευτικά δικαιώματα και όπως πολύ ορθά ανέφερε προηγούμενα ο κύριος Βόποτα ενδιαφέρομαστε όχι μόνο για τη χριστιανική θρησκεία αλλά για τα δικαιώματα όλων των θρησκειών για το δικαίωμα κάποιος να ασκεί την θρησκεία την οποία πιστεύει και πολύ περισσότερο να υπάρχει μια κατανόηση της όλων των θρησκειών και μια κατανόηση της πίστης που έχει κάποιος ως πολίτης. θα ήθελα όμως και λόγω καταγωγής να αναφέρω ένα συγκεκριμένο συμβάν το οποίο έγινε στην κύπρο και αναφέρεται στην έκθεση είναι ότι σε μια εκκλησία που επί δεκαετίες γίνεται η τελετή των χριστουγέννων επί δεκαετίες επενέβη η τουρκική κατοχική παρουσία για να σταματήσει την τέλεση αυτής της λειτουργίας και πολύ περισσότερο να εκδιώξει τους πιστούς και να αναγκάσει τον ιερέα να βγάλει τα ρούχα του. δυστυχώς η διαφοροποίηση αυτού του συγκεκριμένου επεισοδίου είναι ότι γίνεται δυστυχώς δυστυχώς επαναλαμβάνω γίνεται ή ευτυχώς διότι μας δίνεται η δυνατότητα να συνδράμουμε για τη λύση αυτού του προβλήματος σε ευρωπαϊκό έδαφος. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρής τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, η βάρβαρη απόπειρα, η βάρβαρη τρομοκρατική πράξη μάλλον στην Αλεξάνδρη, Αλεξάνδρεια προσθέθηκε σε τόσες άλλες στο Ιράν, στο Πακιστάν. Δηλαδή έχουμε διώξει των χριστιανών, πράγμα το οποίο δεν εμφανίζεται στον τίτλο ε, της πρότασής μας. Θύματα είναι βασικά στη Μέση Ανατολή. Τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των προσδοκιών των 12 εκατομμυρίων χριστιανών που ζουν σε αυτή την περιοχή και που δεν πρέπει ή να μετα... μεταγκαταστούν ή να πεθάνουν. Δεν θέλουμε να στιγματίσουμε μία θρησκεία σε σχέση με μία άλλη, αλλά πρόκειται για φανατικούς Ισλαμιστές που σκοτώνουν την ελευθερία και τους ανθρώπους. Λέιδη Άστον, σας παρακαλώ, τέλος του μηνός στη συνεδρίαση Υπουργών Εξωτερικών να βρεθεί μία απάντηση συντονισμένη σε αυτές τις τρομοκρατικές πράξεις είναι απαραίτητο να ασκήσετε πίεση μέσω των συμφωνιών ε, σύνδεσης με αυτές τις χώρες ώστε οι ένοχοι να μπορέσουν ε, να βρεθούν και να γίνει δίκη τους. Ελευθερία λατρεία σε όλο τον κόσμο λοιπόν είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει να μην πιστεύει. Είναι αυτή η ελευθερία που επιτρέπει τον διαχωρισμό των λατριών αλλά αυτή η ελευθερία αν δεν γίνει σεβαστή κινδυνεύουν όλες οι άλλες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πορέμπα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Lady Άστον. Ε, πολλές από τις θρησκευτικέ διώξεις γίνονται κατά των χριστιανών και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να παραμείνει ανενεργή. Πρέπει να ενεργήσει πραγματικά, να ενεργοποιηθεί. Η συζήτηση που έχουμε σήμερα έχει στόχο να εξασφαλίσει ενότητα στην Ευρώπη, στη δράση κατά της απειλής της θρησκευτική ελευθερίας παγκόσμια. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο μηχανισμό μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποφύγει τέτοια πράγματα μελλοντικά. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να εξασφαλίσουμε η ελευθερία για τη λατρείας να θεωρείται από τα σημαντικότερα ζητήματα στην ατζέντα εξωτερικής πολιτικής. Καθώς υπογράφουμε με τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουμε διατάξεις που να καθιστούν αδύνατη τη θρησκευτική δίωξη. Επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο παρακολούθησης των διώξεων αυτών παγκοσμίως ώστε να έχουμε ενημέρωση για να μπορούμε να, να αντιδράσουμε γρήγορα. Επίσης δεν πρέπει να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Ανοίγουμε τη μετανάστευση από πολλές χώρες, τους επιτρέπουμε να έχουν τόπους λατρείας, αλλά πολύ σπάνια μιλάμε για τους χριστιανούς σε αυτές τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Ε, ε, η ύπαρξη μιας βίβλου μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση ή θάνατο σε αυτές τις χώρες. Είναι αδύνατο να οικοδομηθούν ε, χριστιανικές εκκλησίες σε αυτές τις χώρες. Λοιπόν, πρέπει να επιδιώξουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων των χριστιανών παγκόσμια. Πρέπει να μιλήσουμε δυνατά και στεναρά για την προάσπιση των όλων των θρησκειών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλάν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση εν ώψη των τελευταίων γεγονότων κατά της θρησκευτική ελευθερίας και κατά της ζωής των χριστιανών. Ε, αναφέρομαι ειδικότερα στο Πακιστάν, το Ιράκ, την Ιγυρία και την Αίγυπτο. Το άρθρο 18 της Παγκόσμιας Διακήρυξης αναφέρεται με σαφήνεια στην θρησκευτική ελευθερία. Δυστυχώς, πρόκειται για ένα δικαίωμα που δεν γίνεται πολύ σεβαστό σε πολλές χώρες και το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε δηλαδή ότι η χριστιανική θρησκεία μπορεί να στηγεί τη ζωή του ατόμου. Πρέπει να προασπιστείτε, λέει η Άστον, με σαφήνεια το θρησκευτικό δικαίωμα. Πρέπει να επιδιώξετε την ε, ελευθερία και την ασφάλεια για τη διοκόμενη κοινότητα των χριστιανών. Πρέπει να ε, τιμωρηθούν οι ένοχοι όταν είναι αυτό εφικτό το σήμα αν θέλετε της Ευρώπης είναι η ελευθερία και συμπεριλαμβάνει την ελευθερία λατρείας που είναι η καρδιά της ανθρώπινης ελευθερίας. Είναι και ο δρόμος προς την ειρήνη όπως το ε, είπε ο Πάπας στο μήνυμά του το πρόσφατο. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο χριστιανισμός έχει σχέση και με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Θα ήταν παράδοξο λοιπόν η Ευρώπη να μην ζητά τον σεβασμό των χριστιανικών δικαιωμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ψήφισμα έχει διάφορες, δια... Ε, διάφορες τοποθετήσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων της λατρείας γενικά. Ελπίζω, λέει Διάστον, ότι θα προχωρήσετε δραστήρια και ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα τοποθετηθεί σωστά. Ευχαριστώ, Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα περνάμε στον κύριο Ρέπο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, η αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση Εξωτερική Πολιτική θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο προασπίζει τα βασικά δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανθρώπινα δικαιώματα, κράτο δικαίου, δημοκρατία και ανεξαρτησία. Ε, αυτή τη στιγμή ε, ο πολιτικό νόμο στην ε, Αίγυπτο ανεκαταστάται σιγά σιγά με την Σαρία και από αυτό υποφέρουν κυρίω οι κόπτε. Ο διάλογος χριστιανών και μουαμεθανών είναι μια πολύ παλιά παράδοση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την ευρωπαϊκή πολιτική. Οι χριστιανικές θρησκείες και άλλες θρησκείες είναι κινήματα ειρήνης. Ε, η θρησκεία κανονικά ενώνει τους ανθρώπους, δεν τους χωρίζει. Δεν επιτρέπεται οι τρομοκράτες να χρησιμοποιούν τη θρησκεία σε ένα μέσο βάρβαρης πολιτικής. Ευχαριστώ. Πλωτέρ Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οργάνωση κατά της, ε, ε, της δίωξης για θρησκευτικούς λόγους λέγεται ότι είναι τεράστια ρυθμή ε, των χριστιανών που διώκονται. Τα τελευταία χρόνια 170.000 άνθρωποι πέθαναν επειδή ήταν απλώ και μόνο χριστιανοί. Αυτά είναι τα στοιχεία από μια έκθεση μια οργάνωση που ακριβώς ε, παρακολουθεί τα θέματα των διώξεων των χριστιανών και είναι ξεκάθαρα από τα στοιχεία αυτά ότι είναι η πιο ευάλωτη ομάδα οι χριστιανοί. Η κατάσταση στις Ισλαμικές χώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμη γιατί οι χριστιανοί εκεί θεωρούνται ότι είναι ε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε άνθρωποι να πεθαίνουν απλώ επειδή λατρεύουν ένα διαφορετικό Θεό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει γλίγορα στο θέμα αυτό της δίωξης των χριστιανών που θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο σημαντικό για τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι διώξεις αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε επίσης να θεωρήσει υπεύθυνη τη Βαρόνη ε, Άστρον για να αναλάβει πιο υπεύθυνε ε, ε, δράσεις. Ευχαριστώ. Κύριος Μίτσολ, ένα μισή λεπτό. Καταρχήν, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τη συζήτηση αυτή και το ψήφισμα που υπάρχει. Έχουμε εδώ έναν ε, γίγαντα που κοιμάται ε, γιατί αν αυτή η βία είχε εφαρμοστεί κατά της μουσουλμανικής ε, ε, ε, κοινωνίας θα είχα επίσης εγώ αντιδράσει κατά τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Κύπρο. Η τουρκική κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι τους θεωρούν ότι είναι σωστό οι χριστιανοί να πρέπει να έχουν ειδική άδεια για να ε, λειτουργηθούν και εάν θεωρούν ότι η άδεια αυτή δεν έχει ληφθεί σωστά, να τους βγάζουν έξω από την εκκλησία. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό. Εγώ θα ήθελα να ε, αναφερθώ σε εκείνους τους μαμιθανούς που υποστήριξαν τους Ρουσιανούς σε τέτοιες περιπτώσεις αυτές. Δεν υποστηρίζω και δεν μπορώ να δεχθώ ποτέ βία κατά ατόμων ή κοινωνιών λόγω των, χριστιαν... των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων. Εδώ συζητάμε τώρα για τους χριστιανούς. Πολλοί θεωρούν ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να δεχθούν οτιδήποτε τους κατηγορείται. Αυτό είναι πολύ πεπελειωμένη άποψη. Εγώ σέβομαι εκείνους εδώ στο σώμα που δεν έχουν τις ίδιες θρησκευτικές πεπιθήσεις ή δεν έχουν καμία θρησκευτική πεπιθήση αντίθετα από μένα και που προσπαθούν όμως να υποστηρίξουν τις απόψη μου, γιατί νομίζω διαφοροποιημένοι θα είμαστε ενωμένοι. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ, πρόεδρο, και θα να δώσω το λόγο στην κυρία Κοπά για ένα λεπτό. Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα θρησκευτική βία σε όλο τον κόσμο, γεγονό που προκαλεί ανησυχία και αγανάκτηση. Η απαγόρευση άσκηση τη θρησκευτική πίστη αποτελεί κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και του διεθνού δικαίου, το οποίο ορίζει ότι το δικαίωμα στην πίστη είναι αναφέρετο και δεδομένο η απαγόρευση τέλεσης της λειτουργίας των χριστουγέννων στο ριζοκάρπασο της κατεχόμενης κύπρου από τις δυνάμεις κατοχής οι βομβιστικές επιθέσεις στο χριστιανικό ναό της αλεξάνδρειας εναντίον της κοπτικής κοινότητας είναι δύο μόνο δείγματα της αυξανόμενης έντασης και θρησκευτικού μίσους που αναπτύσσεται σε πολλά μέρη όχι μακρινά από την ευρώπη η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία στην πράξη να περιφρουρήσουν το δικαίωμα κάθε θρησκευτικής πίστης και πρέπει το μήνυμα να είναι ισχυρό και σαφές ότι δεν υπάρχει ανοχή εκ μέρους της ευρωπαϊκής ένωσης σε τέτοια φαινόμενα. θα ήθελα να παρακαλέσω την ύπατη εκπρόσωπο να συμπεριλάβει στις προτεραιότητές της και την αξιολόγηση της κατάστασης της ελευθερίας θρησκευτικής έκφρασης τέλος σε επίπεδο συμβουλίου και ευρωπαϊκής επιτροπής καλό θα ήταν να περιλαμβάνει την πτυχή της προστασίας της θρησκευτικής πίστης σε όλες τις συζητήσεις με τρίτες χώρες. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ε, ήθελα να σας πω το εξής. Η ταυτότητα της Ευρώπης ήταν ε, ένα τμήμα της πάντα η, η χριστιανική θρησκεία. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να παραμένει απαθής όταν εξετάζουμε το θέμα της δίωξης των χριστιανών που είναι μειονότητα στην Ασία, σε Ισλαμικές χώρες και έτσι απειλούνται συνεχώς από δίωξη. Πολλές φορές πεθαίνουν από αυτού του τύπου την βία. Έχουμε διάφορα μέσα στην ε, διάθεσή μας που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τέτοιες πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταδικάζει αυτή του είδους τη βία. Το πιο αποφασιστικό μέσο θα ήταν στις συμφωνίες μας με αυτές τις χώρες να υπάρχει μια ρήτρα η οποία να υποχρεώνει τις χώρες αυτές να φροντίζουν να γίνεται σεβαστή τα τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ευχαριστώ η κυρία Πακ. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητή κυρία Επίτροπε. Το 2009 είχαμε ε, προωθήσει τον διαπολιτιστικό διάλογο στην Ευρώπη. Οι Ορθόδοξοι με τους Καθολικούς, οι Προτεστάντες με τους Ορθόδοξους, οι Χριστιανοί με τους Μωμεθανούς. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε έτσι κάποια κλίματα εμπιστοσύνη. Το κάνουμε αυτό εδώ στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει από ταυτόχρονα ότι έχουμε μια άποψη και θα πρέπει να τολμήσουμε να παραδεχτούμε την άποψη αυτή. Καμιά φορά αυτό είναι λυπές και αυτή τη στιγμή φαίνεται το ίδιο όταν βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε ένα ημερολόγιο για την νεολαία όπου αναφέρονται όλες οι άλλες ε, γιορτές, θρησκευτικές γιορτές εκτός από τις χριστιανικές αυτό θα κάνει μόνο εκείνους που ασκούν βία και διώκουν τους χριστιανούς στην Αίγυπτο να συνεχίσουν οι χώρες που αναφέρθηκαν θα πρέπει να υπογραφούν να βοηθήσουν Ζούνε σε χώρες όταν μιλάμε για την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, το Ιράκ και το Ιράν, σε χώρε λέω από τι οποίε προήρθε η χριστιανική θρησκεία, δεν επιτρέπεται οι άνθρωποι αυτοί να επιτρέψουν να νιαγδοχθούν από τι πατρίτε του. Δεν είναι μειονότητε, είναι Αιγύπτιοι, είναι Παλαιστίνοι, Όπω και όλοι οι άλλοι θέλουν εκεί να ζήσουν και του δυσκολεύουν τη ζωή. Θα πρέπει νομίζω να του υποστηρίξουμε και να προσπαθήσουμε να φροντίσουμε σε όλε τι συνθήκε που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με να αναφέρεται η ανεξιθρησκεία. Να εξασφαλίζεται η ανεξιθρησκεία και να είναι σίγουρο να μην διώκεται κανένα από την πατρίδα του για λόγου θρησκευτικού. Ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ και δίνω τον λόγο στην κυρία Όμενο Ρόουτεν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν βλέπω τις εικόνες από την Βαγδάτη, από την Αλεξάνδρεια, ομολογουμένως μοιάζει σαν να είμαστε μισό αιώνα πίσω. Τότε υπήρχαν θρησκευτικέ διαμάχες μεταξύ προτεσταντών και καθολικών, αλλά αυτά έχουν τελειώσει τελείως για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η Βαγδάτη και η Αλεξάνδρεια ουσιαστικά μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι πρόκειται για μία έκφραση μιας υφέρπουσας κατάστασης σε πολλές χώρες. Γι' αυτό λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου αλλά και μέσα στο πλαίσιο των ελευθεριών μας πρέπει να φροντίσει ώστε σε κάθε συμφωνία, με κάθε μέλος, με κάθε κράτος με το οποίο έχουμε σχέσεις και το έχω προβλέψει για την τουρκική συμφωνία, δηλαδή τον σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών πρέπει να εγγράφεται μια τέτοια διάταξη. Ε, πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα. Το Ισλάμ δεν είναι πλειοψηφική θρησκεία. Θα πρέπει να έχει και αυτή δικαίωμα για ελευθερία. Ωραία όπου είναι μειοψηφική. Πιστεύω ότι η βία που βλέπουμε είναι απαράδεκτη και μαζί μέσω διαλόγου πρέπει να λύσουμε το θέμα. Γι' αυτό σας ζητάω, λέει διάστον να φροντίσετε μαζί με τις υπηρεσίες σας ώστε σε, σε όλες τις χώρες, σε κάθε επαφή που θα έχετε η ελευθερία η θρησκευτική να τίθεται επιτάπητος με τις αρχές. Και στο Ευρωκοινοβούλιο σίγουρα θα βρείτε τη συνεργασία που χρειάζεστε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Η κυρία Θεοχάρου, που τώρα έχει το λόγο εναντίον των χριστιανών στη μέση ανατολή είναι συνήθως έργο φανατικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι διώξει εναντίον των Ελληνοκυπρίων χριστιανών στην κατεχόμενη Κύπρο είναι έργο τακτικού στρατού χώρα που επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω στα χέρια μου επιστολή που έστειλε ο αυτοαποκαλούμενος πρέσβης της τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας κύπρου στις βρυξέλλες μιας οντότητας η οποία υφίσταται μόνο και μόνο στηριζόμενη στην δύναμη του τουρκικού στρατού κατοχής με την οποία επιδιώκει να μεγελιοποιήσει και παράλληλα παραδέχεται ότι η διακοπή της λειτουργίας στο ριζοκάρπασο έγινε διότι οι, χριστιανοί χριστιανοί δεν είχαν βγάλει άδεια Βαρόνι Άστον, από πότε η άσκηση της θρησκευτική πίστης χρειάζεται άδεια από τον οποιοδήποτε και πόσο θα ανέχεστε μια χώρα η οποία επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παραβιάζει τόσο βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικέ ελευθερίες Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε. Δεν είναι παραδεκτό για μας χριστιανοί στη Μέση Ανατολή να υπόκεινται σε τέτοιες επιθέσεις. Ιράκ, Νιγηρία, Πακιστάν. Αυτές είναι χώρες ε, που είχαν χριστιανούς μέσω των αιώνων. Δεν θέλουν να φύγουν οι χριστιανοί πολίτες αυτών των χωρών από τη χώρα τους και είναι πραγματικά λυπηρό που οι Ισλαμιστές συνάδελφοι υποστηρίζουν την αντιχριστιανικές διαθέσεις σε πολλές ομιλίες τους και δηλώσεις τους στο βόρειο Ιράκ. Ε, δεν τολμούν οι άνθρωποι να διακοσμήσουν ανάλογα το σπίτι του αλλού δολοφονούνται άνθρωποι. Ε, συναντηθήκαμε και με επισκόπους από τις περιοχές αυτές και μας ζήτησαν την υποστήριξή μας από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα ώστε οι θρησκευτικέ πεπιθήσεις να μην είναι λόγος θανάτου. Έχουμε την Τουρκία που θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιτρέπει τις ε, θρησκευτικές κοινότητες των χριστιανών. Πού είναι όλοι αυτοί οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ευζοίας των ζώων κτλ. Δεν θα κάνουν κάτι. Τι να κάνουμε τώρα, να δημιουργήσουμε ομάδα για την προστασία των χριστιανών ανά τον κόσμο. Και τώρα περνάμε στον επόμενο ομιλητή τον κύριο Στάστνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είπατε εκπρόσωπε, είναι πολύ ανησυχητικό να έχουμε όλο και περισσότερες επιθέσεις, βίες επιθέσεις κατά των χριστιανών και των κοινοτήτων τους. Όσοι είναι υπεύθυνοι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι είναι φανατικοί, φανατικά ακραία στοιχεία ισλαμικά. Πρόκειται για καθαρό μίσος, πρέπει να σταματήσει, είναι απαραίτητο να σταματήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της και το Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πιέσουν τις κυβερνήσεις όπου εμφανίζονται αυτές οι βίες πράξεις, ιδιαίτερα τις χώρες όπου πραγματικά κάνουν τους τυφλούς, ότι δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Πρέπει εμείς θεωρούμε απαραίτητη κάθε ζωή. Τιμωρούμε όποιον απειλεί την ζωή σε όποια μειονότητα και αν ανήκει το άτομο. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επιμείνουμε και να βοηθήσουμε χώρες να προσφέρουν παρόμοιο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και να τιμωρούνται οι ένοχοι αυτών των απεχθών εγκλημάτων. Εάν δεν γίνει τίποτα θα ενισχυθεί η τάση αυτή. Συνεπώς όλος ο πολιτισμένος κόσμος πρέπει να καταβάλει προσπάθειες να ανατρέψει αυτή την επικίνδυνη τάση. Ευχαριστώ κύριε Στράσιν. Η κυρία Εσάια ε, τώρα για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, Lady Άστον, οι στατιστικές δείχνουν με σαφήνεια ότι 70% όσων απειλούνται ή δολοφονούνται για την θρησκεία τους είναι χριστιανοί και πολλοί χριστιανοί ανά τον κόσμο είναι αντικείμενο βίας. Έχουμε τη Μέση Ανατολή και τα πρόσφατα γεγονότα. Ε, έχουμε τις επιθέσεις κατά θρησκευτικών τελετών στο Ιράκ, στη Συρία, στην Αίγυπτο. Ε, ε, δεκάδες, ανθρώπων δολοφονήθηκαν και παιδιά και στην Ασία Υπάρχουν τεράστιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, στο Βιετνάμ και η ελευθερία ε, ε, λατρείας υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Τα κράτη τα μάτια τους λόγω εμπορικών ε, σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μπορεί να κάνει πάρα πολλά για να βελτιώσει την κατάσταση των χριστιανών ανά τον κόσμο. Βάζοντας μια διάταξη για θρησκευτική ελευθερία σε όλες τις συμφωνίες έχετε μια τέτοια πρόθεση, λέει διάστον. Έχετε την πρόθεση να περιλάβετε μια τέτοια ε, διάταξη και να εφαρμόζετε κιόλα. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί σε μια απώλεια της αξίας των ε, ιδεολογιών μας. Ε, το παράδειγμα της κυρίας Σπακ είναι εκοφαντικό. Ε, οι χριστιανικές γιορτές δεν αναφέρονται στο ημερολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, θα πρέπει και εμείς να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Ο κύριος Μουγκοριάνο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή δεν είναι κάτι το τυχαίο δεν να μιλάμε για ε, λυπηρά γεγονότα, αλλά και μη συντονισμένες ε, επιθέσεις. Πρόκειται για μια κατάσταση μαζικού αφανισμού. Δυστυχώς οι χριστιανοί εκδιώκονται, σκοτώνονται μέσα στα πλαίσια μιας ε, διαδικασίας θρησκευτικής κάθαρσης και τι κάνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να αρκεστούμε σε αυτά και να παρηγορήσουμε τα εκατομμύρια μουσουλμάνους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μέση Ανατολή στην ουσία ακολουθεί μια διαδικασία κάθαρσης. Δεν μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για ελευθερία και ταυτότητα. Ακόμα και εμείς που δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ο χριστιανισμός μια εξωτική και απομακρυσμένη αίρεση, δεν είμαστε έτοιμοι να δούμε αυτή τη μορφή ε, κάθαρσης και παραπλάνησης. Νομίζω ότι η θρησκευτική ελευθερία θα πρέπει να αποτελεί πρόκριμα για τις σχέσεις μας με τα ελεύθερα κράτη και θα πρέπει να εγγραφεί στο νόμο και να αποτελέσει μέρος της εντολής της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Ευχαριστούμε κύριε Ουγκουρεάνο. Ο κύριος Κέλαμ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύρια Ήπατη εκπρόσωπε, σε αυτή την κατάσταση οι δηλώσεις και οι καταδίκες, οι προφορικές δεν αρκούν. Πιστεύω ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι επιθέσεις κατά των χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και τη Νότιο Αφρική και τη Βόρεια Αφρική, με συγχωρείτε. Δεν μπορούν οι χριστιανοί πια να ζήσουν ε, ως μειονότητα και να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις. Δεν μιλάμε πια για νέες μειονότητες, διότι πρόκειται για τους προαιώνιους κατοίκους αυτής της περιοχής. Τώρα εκδιώκονται και πρέπει να φύγουν από αυτές τις χώρες ή γίνονται εσωτερικοί πρόσφυγες, όπως ισχύει και στο Ιράκ. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη θρησκευτική ελευθερία και να ορίσουμε μέτρα κατά αυτών των χωρών που δεν προστατεύουν τις θρησκευτικές μειονότητες. Ο κύριος Ορέχα μίλησε για έναν κατάλογο θυμάτων και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να ε, γνωστοποιήσει αυτό τον κατάλογο. Γιατί μιλάμε για μία πολιτική η οποία είναι εσκεμμένη και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πιο εύκολο να μπορέσει να χτίσει κανείς εκκλησία, είναι πιο δύσκολο να χτίσει κανείς εκκλησία ε, παρά να, να μπορέσει να χτίσει ένα τζαμί στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπουζούτιλ. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις κατά των χριστιανών και είναι πρώτη στο καθήκον μας να αντιδράσουμε. Εάν δεν υπερασπιστούμε με στην Ευρώπη το λίκνο της χριστιανοσύνης, όλες τις μορφές θρησκευτική ελευθερίας, τότε ποιος θα το κάνει στη δική μας θέση. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν δόλοι χειρισμοί των μουσουλμάνων από, ε, να μην γίνουν υποχείριο οι μουσουλμάνοι των εξτρεμιστικών στοιχείων. Κανένας ε, δεν προασπίζει την βία και τις ακραίες αυτές αντιδράσεις. Πιστεύω ότι όλοι οι μουσουλμάνοι θα πρέπει να καταδικάσουν αυτή την τάση. Νομίζω ότι θα πρέπει και οι μουσουλμάνοι να απομακρυνθούν από αυτή την τάση για να προασπίσουν, για να προασπιστούν τον ίδιο το μουσουλμανικό κόσμο. Επίσης, όπου διώκονται οι χριστιανοί θα πρέπει να υπάρξει η σωστή αντιμετώπιση και προστασία των μειονοτήτων αυτών. Πέρα και παρά τα γεγονότα τα οποία ε, ζούμε δεν θα πρέπει να χάσουμε την ε, ε, λογική αυτή. Δηλαδή, το, νομίζω ότι δεν είναι σκόπιμο παρά να ακολουθήσουμε μία φιλιρινική πολιτική, όπως έλεγε και ο Μοχάτ Μακάντι. Ο κύριος Κασίνη, νομίζω ότι οι προλαλήσαντες είπαν ότι έπρεπε να υποθεί. Στην ουσία αποτίμησαν την κατάσταση και προέβησαν σε συγκεκριμένα ε, αιτήματα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να προσθέσω κάτι το οποίο δεν έχει λεχθεί. Ένας μεγάλος Ευρωπαίος, ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, ο οποίος συνεισέφερε στην ε, πτώση του τείχους του Βερολίνου έλεγε ότι οι τέσσερις αξίες που μας διέπουν είναι η ζωή, η ειρήνη, το ψωμί και η θρησκευτική ελευθερία, η ανεξιθρησκεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το τι είχε πει ο ε, ε, δήμαρχος της Φλωρεντίας επί του θέματος. Είπε ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι το μέτρο πρέπει να είναι ο άνθρωπος και μέσα στα πλαίσια ε, της Ευρώπης των αξιών ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο της ε, θρησκευτικής ενότητας. Θα πρέπει να μπορεί να συνομιλεί με το Θεό και αυτό που έχει σημασία είναι να μην αρνούμαστε την ε, ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Θεωρώ ότι αυτές οι σκέψεις θα μας βοηθήσουν και θα βοηθήσουν και την ύπατη εκπρόσωπο να μπορέσει να διαμορφώσει μία σκέψη η οποία να προασπίζει τα δικαιώματα του ανθρώπου και, και, ε, και να προασπίζει και την ε, ανεξιθρησκεία. Λοιπόν, στη διαδικασία Catch the Eye υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα διότι έχουμε 20 υποψήφιους ομιλητές και έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να λάβετε το λόγο, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Ο κύριος Αλάμα έχει το λόγο. Εγώ θα περιοριστώ στο εξή. Θα ήθελα η ύπατη εκπρόσωπος, κυρία Άστον, να εντάξει στην ατζέντα των σχέσεων με την Αίγυπτο και ένα ειδικό θέμα. Δηλαδή, να ζητήσουμε από τις Αιγυπτιακές αρχές να βγάλουν από τα επίσημα έγγραφα, από τις ταυτότητες, τα διαβατήρια, και όλα τα έγγραφα εργασίας στην ε, μνήα στο θρήσκευμα, διότι στην ουσία υφίστανται οι χριστιανοί διακρίσεις τη στιγμή που στο ε, επίσημο έγγραφό τους αναγράφεται το θρήσκευμά τους. Σήμερα η μουσουλμανική τρομοκρατία εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία διάκρισης κατά των ε, χριστιανών που θεσμοθετείται. Αυτό είναι ένα άμεσο αίτημα διότι αν δεν γίνεται αυτή η ρητή μνήμα, τότε δεν θα υπάρχει θεσμική τρομοκρατία. Η προς Ευχαριστώ. Η κυρία Παπαδοπούλου. Mr. President, Articles 3 and... Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 3 και 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απαγορεύει την απάνθρωπη ή ε, ταπεινωτική συμπεριφορά και αναφέρεται στο δικαίωμα της ανεξιθυσίας. Αυτό επανελήφθη πλειστάξει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην απόφαση του της υπόθεσης του Κύπρος κατά της Τουρκίας το 2001. Λέει διάστον, δυστυχώ για τα τελευταία 36 ε, χρόνια η Τουρκία, μια χώρα υποψήφια για την ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστρέφει θρησκευτικά μνημεία στην Κύπρο, <clears throat> διώκει τους χριστιανούς, και τέλος, απαγόρευσε ε, τον φώτων την ε, λειτουργία στην Βόρξο και στο Διαλούσα. Θα πρέπει να καταδικαστεί η Τουρκία για τα εγκλήματα αυτά στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να μείνει απαθής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειλούνται οι χριστιανοί στην Κύπρο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τράιν, παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ψήφισμα για την κατάσταση των χριστιανών παγκόσμια σχέση με την εξεθρησία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών ανά τον κόσμο οι φιλελεύθεροι είναι εκείνοι που προωθούν εδώ το θέμα και αυτό μας κάνει να διαφοροποιούμε από τους συντηρητικού που αναφέρονται μόνο στο θέμα των χριστιανών γιατί δεν πρόκειται για θέμα μόνο των χριστιανών από φιλελεύθερη σκοπιά πρόκειται για θέματα ανεξαιρεσίας γενικά όλες τις θρησκείες δηλαδή ανά τον κόσμο πρόκειται για το θέμα της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων και την υποχρέωση κάθε χώρα να προστατεύει τις απειλούμενες θρησκευτικές μειονότητες όπως μπορεί. Και στην Ευρώπη έχουμε προβλήματα. Εγώ είμαι από το Βερολίνο και στην κατάσταση που έχουμε στη Βερολίνο αυτή τη στιγμή ε, είδαμε να υπάρχουν έξι μπριστικές επιθέσεις κατά ε, τζαμιών στο Βερολίνο. Ευτυχώς χωρίς ε, θύματα. Α, προσπαθούμε όμως να προσπαθήσουμε την να προασπίσουμε τα δικαιώματα των μειονοτήτων αυτών. Βέβαια δεν μπορούν να υπάρχει κάτω από, μπροστά από κάθε εκκλησία και τζαμί ένας αστυνομικό, αλλά είμαι κατά της διάθεσης αυτή. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς ως πολιτικοί να αναλάβουμε την ευθύνη για την ατμόσφαιρα που υπάρχει στη χώρα μας κατά των ε, θρηστικών μετεωροθήτων και να είμαστε ε, υπεύθυνοι για την ανοιχτή στάση έναντι όλων των θρησκειών στις χώρες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό έπρεπε να είχατε μιλήσει, όχι ενάμιση. Ο κύριος Στάνοκ. Όταν πρώτο εκλέγηνε εδώ στο σώμα πριν από 11 χρόνια, να κάπως ε, πολύ μυστήριο στο ΕΛΚ γιατί συχνά έθεσα το θέμα της δίωξης ε, των, των διωγμών των χριστιανών Στι ε, μαθηματικές ε, Εν τω μεταξύ τα θέματα επιδεινώθηκαν και γι' αυτό βλέπω ότι ε, και πολλές και από τις αντι δυνάμει δυνάμεις του σώματος ξύπνησαν επιτέλους και είδαν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Το περασμένο Σάββατο ήμουνα μπροστά στην ε, Downing Street αριθμό 10 στο Λονδίνο μαζί με τους κόπτες εκλογισμού για να επίσης το θέμα. Σήμερα ε, καλώ εσάς λέει Διάστον, σαν το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσπίσει επίσης τα θέματα αυτά. Ο κ. Σαλαφράκος έχει το θέμα. Πριν από καιρό είχα γράψει έναν άρθρο με τον τίτλο «Πληθυντικός μονόλογος». Πληθυντικό σημαίνει ότι μιλάμε πολύ και μονόλογο σημαίνει ότι μιλάει ένας. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα των κοινωνιών μας σήμερα. Μιλάμε όλοι και μάλιστα τις περισσότερες φορές για ιδέες και ακούμε μόνο αυτά που λέμε εμείς. Εκεί εντάσσω λοιπόν το πρόβλημα της εξάρσεως του Ισλαμικού φανατισμού που παρουσιάζεται τις ημέρες αυτές, που παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο τις Άγιες Μέρες της Πρωτοχρονιάς. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μέσα σε έναν αιώνα από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τώρα ενώ στην Ανατολή οι χριστιανοί εκπροσωπούσαν το 22% του πληθυσμού τώρα εκτιμούνται σε λιγότερους από 10%. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτή την έξαρση του Ισλαμισμού διότι έχουμε γερασμένες ηγεσίες τόσο στην Αίγυπτο όσο και στη λιβύη όσο και σε άλλες χώρες που δεν ξέρουμε μετά την πτώση τους τι μπορεί να συμβεί και πού μπορεί να οδηγηθούν οι χώρες αυτές. με τα δεδομένα αυτά παρακαλώ κυρία άστον μέσω της επιρροής σας να λάβετε πρωτοβουλίες ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση του θρησκευτικού φανατισμού με ε, αντιστοιχεία και των χριστιανών και των μουσουλμάνων. ευχαριστώ πάρα πολύ. Herr Präsident, der Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ΚΟΠ της Επισκόπος Δαμιών προώθησε πρόσφατα την θρησκευτική ένωση ε, και, μεταξύ χριστιανών και και, Ισλαμισ... και μομεθενών στην Αίγυπτο λόγω των επιθέσεων και στα τζαμιά και στις χριστιανικές εκκλησίες. Όταν σήμερα όμως δείχνουμε να μας ε, έχουμε πληγή δεν πρέπει να απορούμε γιατί από την κεφαλή βρωμάει το ψάρι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και όταν βλέπουμε ότι η Κομισιόν παραδειγματικά εκδίδει ένα ημερολόγιο που διαμείνεται σε 21.000 ε, ε, Ευρωπαϊκό Σχολείο για 3 εκατομμύρια μαθητές που δεν αναφέρονται καθόλου θρησκευτικές χριστιανικές γιορτές αλλά ινδουιστικές, βουδιστικές και άλλες αυτό τι σημαίνει εμείς πρέπει να είμαστε ε, σωστοί και να μην δεχθούμε καθόλου την ανοχή Ευχαριστώ κυρία Ζαβόσκα έχει το λόγο Ευχαριστώ πρόεδρε Κυρία Άστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή μετά από την δίωξη των ε, χριστιανών τη στιγμή που έχουν εκδιωχθεί από τις οικίες τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να τύχουν προστασία οι χριστιανοί. Και η προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένη. Πιστεύω ότι αυτή η ιδεολογία καταπατά την ανεξιθρησκεία και οι χριστιανοί θα πρέπει να τύχουν καλύτερης προστασίας. Πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν προβλήματα την ε, παρουσία θρησκευτικών εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις θανατηφόρες ε, επιθέσεις όπου σκοτώθηκε και ένας αρχιεπίσκοπος και πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη Βιέννη υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την καταπολέμηση της, ε, της ε, καταπάτησης αυτών των δικαιωμάτων των χριστιανών. Τέκης. Ε, Ως ε, μέλος μίας μειονότητας στη Ρουμανία ήξερα πολύ καλά τις διώξεις επί Τσαουσέσκου όταν ζήσαμε αυτό τις, αυτές τις διώξεις του. Ο Βίκτορ Ορμπάν έθεσε ως προτεραιότητα την καταπολέμηση των διωγμών κατά των χριστιανών. Ελπίζω να μπορέσει λέει, Λέδη Άστον να συνεργαστεί με την Ουγγρική Προεδρία στην Ισταμπούλ. Είδαμε μεγάλες διώξεις Αρμενίων και Ελλήνων που σκοτώθηκαν, διώχθηκαν κατά τον 20ο αιώνα και βλέπουμε μεγάλους διώγμους χριστιανών. Νομίζω ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων μαζί με την κυρία Χάουταλα θα πρέπει να θέσει αυτό το θέμα επιτάπητος και θα ήθελα στις 31 Ιανουαρίου, ε, κυρία Άστον, κατά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα, διότι αυτή είναι μία από τις ε, προτεραιότητες. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους χριστιανούς. Και τώρα δίνω το λόγο στη Lady Ashton. Για να τελειώσουμε με τη συζήτηση αυτή και για να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία θέματα από τις πολλές ιδέες που έχουν προταθεί. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους αντιλαμβάνομαι πόσο έντονα είναι τα αισθήματά σας και πόσο προσπαθείτε να στηρίξετε το έργο μας σε αυτό το τομέα. Όπως έλεγα, ένας λόγος που αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένη να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι έχει τεθεί το θέμα και ε, στο Συμβούλιο και θα επανέλθουμε στο τέλος Ιανουαρίου. Τα σχόλιά σας ε, απηχούν αν θέλετε ε, τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί προς εμένα και από υπουργού και από κράτη που ανησυχούν. Θέλω να αποσαφηνίσω ότι πράγματι μίλησα για τη χριστιανοσύνη. Διατύπωσα τους λόγους για τους οποίους πήγα στη Βιθλεέμ. Το έπραξα αυτό για να αναγνωρίσω ότι αν και βρισκόμουν στη Μέση Ανατολή στην καρδιά πολλών θρησκειών την παραμονή των χριστιανικών Χριστουγέννων ήταν πολύ συγκεκριμένη η παρέμβασή μου. Δυστυχώς ο κ. Λάγκας δεν είναι πλέον στη του για να με ακούσει αλλά πράγματι πιστέψτε με έκανα αυτή τη δήλωση στην Πεθλέα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά θέματα που θίξατε. Πολύ αναφερθήκατε στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που είναι στη διάθεσή μας ώστε να εξασφαλίσουμε την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μέσα στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών που έχουμε συνάψει από το 1995 έχουμε περιλάβει μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υφίσταται αυτή η διάταξη στις συμφωνίες με 134 χώρες. Ο βασικός λόγος είναι να υπάρξει αμοιβαία δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι και η νομική βάση κυρώσεων σε περίπτωση που έχουμε σοβαρές παραβιάσεις. Θα θυμόσαστε ότι κατά το παρελθόν με άλλη ιδιότητα είχα μιλήσει για τη Σρι Λάνκα πολύ και είχαμε λάβει και μέτρα αναστολής λόγω παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξετάζουμε πάντοτε τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας και τον τρόπο που συνάπτουμε συμφωνίες. Ένα από τα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέρον καθώς η Κομισιόν θα εξετάζει το μέλλον του κανονισμού GSP είναι κατά πόσο η επικύρωση συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να περιληφθεί. Τώρα υπάρχει και άλλη πλευρά βεβαίως. Υπάρχουν οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούμε για να υποστηρίξουμε την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υποστηρίζουμε όπως γνωρίζετε προγράμματα για την καταμολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας ε, των διακρίσεων ε, σε κάπου 60 χώρες. Συνεπώς, η ισορροπία μεταξύ των εργαλείων που είναι στη διάθεσή μας είναι σημαντική. Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταδείξουμε ε, την αντίδρασή μας όταν υπάρχει μια σημαντική παραβίαση. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να υποστηρίξουμε και τις ΜΚΟ που είναι πολύ δραστήριες στον τομέα του ρατσισμού και κατά των διακρίσεων γενικότερα. Τώρα, θα ήθελα να μιλήσω για το ρόλο των αντιπροσωπιών μας σε όλο τον κόσμο. Είπα ήδη ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε τα ζητήματα αυτά σε ολόκληρο τον κόσμο και μου έκανε πολύ εντύπωση ε, που πολλοί βουλευτές αναφερθήκανε σε αυτό το οποίο έχει γίνει πολύ πιο αναγνωρίσιμο πρόσφατα, αλλά που ήταν πολύ μεγάλη ανησυχία κατά το παρελθόν. Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο οι οι ιερείς οποιασδήποτε θρησκείας υφίστανται διώξεις σε όλον τον κόσμο πρέπει να τα παρακολουθούμε με βεβαίως αυτά τα ζητήματα όχι μόνο όταν γίνονται βία όταν γίνονται βία είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε αλλά και πριν πρέπει να τα παρακολουθούμε γιατί είναι σπάγια πηγή διακρίσεων συνεπώς πιστεύω ότι οι αντιπροσωπείες μας στο όλο το κόσμο ε, πρέπει να είναι πηγή που μας κοινοποιεί και μας ενημερώνει περιπτώσεις διακρίσεων αν θέλετε είναι οι πρώτες φουσκάλες κάτω από την επιφάνεια που πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη. Μέσα στο πλαίσιο της δουλειά μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα στο πλαίσιο της έκθεσης που θα υποβάλουμε ε, θα αναφερθούμε και στις θρησκευτικέ μειονότητες. Ε, Βεβαίω μιλήσαμε πολύ για τον χριστιανισμό σήμερα, αλλά πολύ σωστά πολλοί βουλευτέ αναφέρθηκαν ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό και ανοχή και για τις άλλες λατρείες. Και θα πρέπει πραγματικά να αντιληφθούμε τι διαδραματίζεται και μέσω των εκθέσεών μας και μέσω των αντιπροσωπιών μας όλο τον κόσμο. Έτσι θα γνωρίζουμε καλύτερα πώς να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που είναι στη διάθεσή μας, ιδιαίτερα από την πλευρά της Κομισιόν. Ταυτόχρονα χρειάζεται και πολιτική θέληση, όχι μόνο ακ μέρους μου, αλλά εσείς σαν κοινοβουλευτικοί έχετε ισχυρή φωνή και μαζί με τα κράτη-μέλη και τους υπουργούς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα πράγματα. Ξεκίνησα λέγοντας ότι δεσμεύομαι να εξασφαλίσω ότι θα βελτιώσουμε τα πράγματα, θα παρακολουθήσουμε τα πράγματα και θα χρησιμοποιήσουμε πολιτικούς και άλλους μηχανισμούς για να διατηρήσουμε αυτό το θέμα ανοιχτό ε, και στο μέλλον. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλιά σας, δεν απάντησα σε όλα. Πήρα όμως σημειώσεις, θα τα σκεφτώ όλα και αυτό θα μας βοηθήσει στη συζήτηση που θα έχουμε στο Συμβουλίο Εξωτερικών Υποθέσεων τέλη Ιανουαρίου. Ευχαριστώ κυρία Άστον, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε λάβει 7 προτάσεις. Και η ψηφοφορία θα γίνει